Uh, <clears throat> κυρίες και κύριοι, Σα ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση και τους ε, ακροατές μας στο διαδίκτυο και από αυτούς το συγγνώμη γιατί αργήσαμε λιγάκι, αλλά έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική πρόταση και αυτό σημαίνει και κάποιες τελευταίες συνεννοήσεις, συνεννοήσεις τελευταία στιγμής, ώστε ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια στεναρή <clears throat> κοινή για αυτές τις τόσο σημαντικές προτάσεις. Σας καλωσορίζω λοιπόν θερμά, είτε εδώ είτε στο διαδίκτυο στην ειδική αυτή σύνοδο της Επιτροπής μας που θα ψηφίσουμε τρεις εκθέσεις από την κυρία Καλνιέτε, τον κύριο Κούρα και τον κύριο Μπουζόη για σημαντικά κεφάλαια της εσωτερικής αγοράς. Προτάση της Κομισιόν. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ψηφοφορία γιατί πιστεύουμε θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε σημαντικές προτάσεις όπως έχει ζητήσει και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας και ο Λουί Γκρέχ ο οποίος είχε διατυπώσει την πρώτη έκθεση προς την κατεύθυνση αυτή είναι εδώ παρόν και τώρα προχωρούμε ένα βήμα περισσότερο από την αρχική του πρόταση και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. <clears throat> Πρωτού ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Σας υπενθυμίζω ότι πρέπει να έχετε τις κάρτες ψηφοφορίες σας. Κάποιοι περιμένουν να έρθουν ακόμα για να τις χρησιμοποιήσουμε. Και λέω στις πολιτικές ομάδες επίσης, όταν έχετε αναπληρωματικά μέλη που δεν είναι κανονικά μέλη, αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής μας, πρέπει να δώσετε, μια, ε, να δώσετε ένα υπόμνημα στο, στη γραμματεία να πληροφορήσετε τη γραμματεία ποιο ψηφίζει στη θέση ποιου. Παρακαλώ δώστε μα ένα σημείωμα εάν δεν το έχετε πράξει ήδη για τα θέματα αυτά. Αυτά για τι επίσημε ανακοινώσει, <coughs> Έχετε το σχέδιο ημερήσια διάταξη. Φαντάζομαι ότι θέλετε να το εγκρίνετε, γιατί το μόνο θέμα που έχουμε είναι η ψηφοφορία. Επίσημη ανακοίνωση επίση. Όσοι από εσά εργάζεστε για την νομοδότηση για την έκθεση Ευρωπαϊκή Ένωση Ανδώρα, έχει αναβληθεί η ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα γιατί η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή εξετάζει ορισμένα νομικά θέματα που συνάπτονται με αυτή τη γνωμοδότηση. Σας λέω και πάλι ότι μεταδίδεται και στο διαδίκτυο αυτή η συνεδρίαση και έχουμε το δελτάριο τα νέα της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ που έχουν διανεμηθεί σε όλα τα μέλη μας και όποιος θα ήθελε να έχει ένα αντίτυπο μπορεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα μας και να γίνει φίλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Έχουμε κάπου 1.500 φίλους που είναι συνδρομητές σε αυτό το, ε, το έντυπο, τα νέα της ΣΥΜΚΟ και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στις 2.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Ψηφίσουμε τώρα. Μία πρόταση να σας κάνω ως εξής. Λόγω του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αυτών των εκθέσεων, επειδή έχουμε πολλές τροπολογίες, προσπαθήσαμε να τις ε, συνενώσουμε ώστε να αναφέρονται στα διάφορα κεφάλαια της ε, έκθεσης και έχουμε και τις γνωμοδοτήσεις από αρμόδιες επιτροπές. Λόγω του ολοκληρωμένου όμως χαρακτήρα αυτής της ε, έκθεσης θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε την τελική ψηφοφορία και των τριών εκθέσεων στο τέλος και μόνο. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες, <clears throat> αλλά όχι την τελική ψηφοφορία για τις, πιο, για τις πρώτες δύο εκθέσεις και μόνο στο τέλος θα κάνουμε την τελική ψηφοφορία και φυσικά οι πολιτικές ομάδες θα εξασφαλίσουν ότι έχουν μια συνεκτική γραμμή για τις τρεις εκθέσεις ομού. Εάν λοιπόν δεν έχετε αντίρρηση, ούτως απεφασίστε. Τώρα, πρωτού ξεκινήσουμε, να ελέγξουμε ότι λειτουργεί το σύστημα ψηφοφορίας και να δούμε τους αριθμούς των βουλευτών που ψηφίζουν. Καταρχήν, μόνο τα μέλη του ΕΛΚ παρακαλούνται να ψηφίσουν. Άρχεται η ψηφοφορία για το ΕΛΚ. Vote is open for the EPP. The vote is closed for the e για το ΕΛΚ. 15 υπέρ μια αποχή. Ωραία αλλά έχετε μόνο 14 μέλη που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Δύο από εσά δεν μπορούν να ψηφίσουν από εδώ και πέρα. Α, κρατήσατε θέση αποχή. Εσεί φταίτε. Κυρία Στάλερ είχε κρατήσει θέση αποχή. Ένα άτομο λιγότερο λοιπόν για το ΕΛΚ πρέπει να ψηφίζει. 14 ψήφοι αντιστοιχούν στο ΕΛΚ εδώ. Να επαναλάβουν την ψηφοφορία. Και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία για τα μέλη του ΕΛΚ και μόνο. Μόνο ΕΛΚ. Τώρα έχετε 13 μέλη που ψηφίζουν μονάχα. Ωραία, 14. Ίσως αν δεν ψηφίσει η συγγήτριά σας μπορεί να συγκεντρωθεί και να σας δίνει τα καλύτερα σινιάλα. Λοιπόν, εντάξει για το ΕΛΚ. Κλείνει την ψηφοφορία. Αρχίζουμε για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τους σοσιαλιστές. Δέκα πρέπει να έχετε, όχι έντεκα όπως έχετε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, εξασφαλίστε ότι θα είσαστε 10 μονάχα. Πέρα στις ψηφοφορίες. Φιλελεύθεροι τώρα. Τέσσερι, εντάξει. <clears throat> πράσινοι. του βλέπω, του βλέπω τώρα. Τρεις, πράσινοι. Τρει συντηρητικοί. Δύο από την ΚΟΕ και ο κύριο Σαββίνη. Ωραία. Εντάξει, είμαστε όλοι παρόντε. Δεν έχουμε μία σου. Προχωράμε. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση Καλνιέτ. Έκθεσης Καλνιέτε, θέλετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις κυρία Καλνιέτε πρώτο ξεκινήσουμε. Έχετε το λόγο. Ναι βεβαίως. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιοδησίτες. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία που κατέληξε σε 17 συμβιβαστικές ε, τροπολογίες επειδή όλοι έδειξαν ένα ανοιχτό πνεύμα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου για τις δύο άλλες εκθέσεις, γιατί συμφωνήσαμε σε μια κοινή δομή στις εκθέσεις αυτές, ώστε να μπορέσουμε να καταδείξουμε και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των προτάσεων για την εσωτερική αγορά fait, Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, σας λέει η συγγήτρια. Αυτά είναι ωραίες στιγμές που δεν γίνονται πολύ συχνά. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό το θαυμάσιο έργο δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς την υποστήριξη της γραμματείας και θέλω να ευχαριστήσω την Καντζόμπα και τον Τάιρον Κούλα για την πολύ καλή του εργασία και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συμβούλους και συνεργάτες από το ΕΛΚ και φυσικά και τον συντονιστή μας τον Ανδρέα Σουάμπ. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Μάλκολμ Χάρμπορ γιατί ως πρόεδρος έχει καταφέρει να συντονίσει τη δράση μας με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. <clears throat> Το σημαντικό τώρα είναι να φτάσει η ενιαία αγορά να είναι μία από τις προτεραιότητες, τις πρώτες προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και την οικονομική διακυβέρνηση. Και προσβλέπω στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ όλους που φέρατε τις εκθέσεις αυτές στο τελικό του στάδιο. Ευχαριστώ, Σάντρα. Και συμφωνώ και εγώ, νομίζω ότι η επιτυχία αυτών των εκθέσεων δείχνει την ικανότητα της Επιτροπής μας να λειτουργεί σε διαπαραταξιακή βάση για ένα τόσο δύσκολο θέμα. Πάμε. Ψηφοφορία. Παράγραφος 1. Τροπολογία της Νομικής Επιτροπής Παριθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 9. Των Πρασίνων. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η εννέα, λοιπόν προστίθεται ως νέα τροπολογία. Επιτροπή Απασχόληση τροποποίηση, Τροπολογία 1 καλύπτεται από την 3 και έχουμε μία σειρά την 11 και 12 θα ψηφίσουμε αργότερα. Πηγαίνουμε στην 13 Τριανταφυλλίδη Σφένσον. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λίγο πιο ναι. γρήγορα αν μπορείτε. Ναι. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 υπέρ, 20 κατά. Ναι. Λίγο πιο γρήγορα αν μπορείτε να ψηφίσετε για να τελειώσουμε κάποια στιγμή. Τροπολογία. 14 καλύπτεται. 16 <clears throat> Μακλάρκιν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Ηλεκτρονικά. πέρας. Απορρίπτεται. <clears throat> Τροπολογία 18 καλλιέται. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτή. παράφος 3, τροπολογία 19 <clears throat> των πρασίνων, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 17-19. Έξι της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Δεν διάβαζα προσεκτικά. Εκπίπτει η 6. Ψηφίζουμε την 5 ε, της απασχόλησης. Ψήφι υπέρ, κατά δεκτή. Οικονομική Επιτροπή 16. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται λογω οψηφιας ισοψηφίας 18-18. Απασχόληση οικονομική 20. Ψήφι κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 20 της εισηγήτριας υπέρ κατά δεκτή. 21 τριανταφυλλίδη. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας απορρίπτεται. <clears throat> Τροπολογία 22, Μήτρο Ρέπο, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Απασχόληση 2, υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβαστική τροπολογία 1, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. <clears throat> μας φέρει αυτό στην παράγραφο 15, Λάκενγκάρ, <clears throat> ως προσθήκη στην παράγραφο 5, ψήφι υπέρ. Κατά, δεκτή. Ένα της Περιφερειακής Επιτροπής υπέρ, καλύτερα ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία Περιφερειακή 1, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 59 γκρέχ. Αρχίζει ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεν σας λέω τα στοιχεία, τα, τα βλέπετε στην οθόνη. Καλύπτεται η επόμενη τροπολογία της ε, Περιφερειακής Επιτροπής. Πάμε στην παράγραφο 6 δεν θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες 25 και 26 γιατί εκπίπτουν με την τροπολογία της Περιφερειακής Επιτροπής παράγραφος 6α το αντίστοιχο κομμάτι της τροπολογίας της Περιφερειακής ψήφι υπέρ κατά δεκτή η νομική επιτροπή τροπολογία 30 ψήφι υπέρ κατά δεκτή εκπίπτει η 18 της απασχόλησης και 18 της περιφερειακής επίσης εκπίπτουν. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχές δεκτή. Εκπίπτει 118. Πάμε στη συμβιβαστική τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 τώρα. Βανιού τη κυρία Βεργιό, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία Πέρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 20-17. Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, το αντίστοιχο κομμάτι, ψήφι υπέρ, ηλεκτρονικά. Στην 3 PC1. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά μονάχα, διαφορά μονάχα. Τροπολογία 34 σε λογά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 19-18. τροπολογία 126 εκπίπτει. Η 37 έχει καλυφθεί. Βλέπετε ποιες έχουν καλυφθεί. Πάμε στην απασχόληση 14. Αυτή την ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Με μία ψηφοδιαφορά μονάχα. Τη εισηγήτριας παριθμών 28 ψήφι υπέρ κατά εγκρίνεται. Οι 12 τη συνομική και οι λίμπε 4 καλύπτονται, οι 39 καλύπτονται, συμβαστή 4 τώρα ψήφι υπέρ. Κατά δεκτή. 9 τη νομική επιτροπή Ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται 10 της νομικής υπέρ κατά επίσης δεκτή 2 της ίντα ψήφι υπέρ ηλεκτρονικά καλύτερα Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2 άρχεται η ψηφοφορία πέρας Απολύπτεται. Η τρία της απασχόλησης δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Είμαστε στη συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Νομική 16. Ως προστίκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 50 σουλιακή άλλων υπέρ κατά δεκτή. Εκπίπτει η δέκα της απασχόλησης και 177 επίσης. Πάμε στην απασχόληση 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Απασχόληση 16. Πέρας. Απορρίπτεται. 51 δεν ψηφίζεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περιφερειακή 17. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Η 58 εκπίπτει. Απασχόληση 11. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 76 Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεχτεί. Πάμε στην 8 των δημοσίων ελευθεριών. Άρχεται η ψηφοφορία, λίμπε 8. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 75 βαζιέρδα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 75. Πέρας. Απορρίπτεται. 77 κρότσμα και 8 απασχόληση. Ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. Λίμπε 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Νομική 12. Άρχεται. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 80. Μακλάρκιν. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 81. Σιάντε Μόζε. Άρχεται. Πέρασε εγκρίθηκε. 22-15. 83 διαγραφής 30 φιλίδι υπέρ κατά απορρίπτεται 84 υπέρ κατά εγκρίνεται 86 των πρασίνων υπέρ κατά εγκρίνεται Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 92 τριανταφυλλίδης. Αυτή την ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Απασχόληση 12. Άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 94. Το αντίστοιχο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Εντ 178. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 22-14. Νομική 14, νομική 4, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Εκπίπτει η τροπολογία του κ. Ρέπο. Λαϊνιόγκοκ επίσης και 91 πηγαίνουμε στην 14 οικονομική. 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 78 εκπίπτει, 98 επίσης, 99. μακλάκι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δημόσιες ελευθερίες 11. Άρχεται και τη Λίμπε 11. Πέρα Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά μονάχα. 197 Βαντεκάμπ. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 100 των πρασίνων. Άρχεται ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 101. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 102. χαρά. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 103 απεσύρθη, 105 δεν ψηφίζεται. Πάμε στην 79. 30 φιλίδες και λεπά. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 106 της εισηγήτριας, υπέρ, κατά, Δεχτεί. Συμβαστική 12. Υπέρ, κατά, Δεχτεί. Συμβαστική 13, υπέρ, κατά εκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά εγκρίνεται Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά εγκρίνεται. 123 καλνιέται μαζί με την 85 από εκείνο ψηφίζονται αυτά υπέρ κατά εγκρίθηκε 1.24 Μπουσουτήλ άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 των αναφορών ως προσθήκη. Ηλεκτρονικά. Petitions 6. Πέρας. Εγκρίνεται. 20-17. 125 έχει αποσυρθεί, 126 και 82 καλνιέται. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Πάμε στην 127 ρέπο. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 1.33 ρέπο. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. 132 εκπίπτει. Και 134 επίσης εκπίπτει. Αιτιολογικές αναφορές. Τροπολογία 1. Τόγια Ταραμπέλα. Άρχεται η ψυχοφορία ηλεκτρονικά για την 1. Πέρασε. Απορρίπτεται. 2 ρεκόρ υπέρ κατά δεκτή αιτιολογικές σκέψεις τροπολογία 3 υπέρ κατά δεκτή 4 De Jong Άρτη την ψηφοφορία 4 πέρας εγκρίνεται 23-14 5 γκρέχ. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 19, 18, 6 των πρασίνων. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 7 δεν ψηφίζεται. Η 8 τώρα. Η 11 και η 32 από κοινού. Αρχίζει η ψηφοφορία για αυτό το μπλοκ. Πέρασε. Απορρίπτονται. Οπότε κλείνουμε με τις τροπολογίες, θα επανέλθουμε φυσικά στην τελική ψηφοφορία, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω για την τόσο καλά προετοιμασμένη ψηφοφορία και τις πολύ καλές συμβαστικές. Περνάμε τώρα στην έκθεση του καθηγητού Αντωνίου Φερνάντο Κορέγια και Ντεκάμπος. Καθίστε παρακαλώ ξανά γιατί έχουμε ακόμη πολλές ψηφοφορίες. Λοιπόν, ησυχία παρακαλώ. Πρώτα θα ακούσουμε τον εισηγητή να μας κάνει μια εισηγησούλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους Κιώδης και όλους τους συναδέλφους γενικά που συνεισέφεραν στην συγγραφή της έκθεσης αυτής. Πετύχαμε 17 συμβιβασμούς Έχουμε ακόμη τρεις εκκρεμούντες. Η παραπομπή στην κοινωνική πολιτική, δηλαδή στην κοινωνική ρήτρα που λένε άλλοι, είναι το αμφιλεγόμενο θέμα. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έκαναν συνάδελφοι από διάφορες ομάδες acceptable at least at αλλά δεν προλάβαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και από αυτό. Πρόκειται βέβαια για μια απλή εφαρμοστική ρήτρα με τους ίδιους όρους που λέμε και στο 29. Η δημόσια διαβούλευση που ζήτησε η Κομισιόν στην πρώτη αναθεώρηση λέει εδώ στην τροπολογία 29 ότι είναι η τέταρτη σημαντικότερη μεταξύ 40 ετούντων πρώτο αίτημα των συνδικαλιστών κλπ. Για μας δεν είναι αποδεκτό λοιπόν η κοινωνική αυτή ρήτρα να μην μπορεί να εγκριθεί. Ιδιαίτερα εφόσον αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικά τα σχόλια των όσων έχουν σχολιάσει αυτή την πρόταση της Επιτροπής. Και δεύτερη διαφωνία είναι για τις υπηρεσίες κοινή ωφελία. Μία φράση είναι όλη η διαφωνία. Εμείς θεωρούμε ότι επειδή συμφωνούν όλοι ότι οι κοινωνικές αυτές υπηρεσίες κοινή ωφελία πρέπει να είναι το τομεακού χαρακτήρα και να είναι τα κράτη αρμόδια. Αλλά χρειάζεται κάποια νομοθεσία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς την οποία θα παραμένει μια νομική αβεβαιότητα και ασάφεια την οποία θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτό είναι ο μόνος λόγος της διαφωνίας λοιπόν. Σας αναφέρω αυτές τις διαφωνίες, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αδύνατο να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Προς στιγμήν όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε τις διαφορές που εκφράζονται εδώ με το αρχικό κείμενο. Θα καταθέσουμε προφορική τροπολογία λοιπόν για ένα τουλάχιστον από τα δύο αυτά θέματα και ελπίζουμε μέχρι το τέλος να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία γιατί θα ήταν κρίμα να παραμείνει εφόσον επί όλων των υπολείπων συμφωνούν όλοι. Καλά, σας ευχαριστώ καταρχήν για το ρόλο που παίξατε, τον ηγετικό ρόλο. Ήμουν και εγώ εισηγητή σε παρόμοιο θέμα και γνωρίζω τις δυσκολίες. Ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όπως έγινε και για την έκθεση Γκρέκ. Σας υπενθυμίζω ότι αν δεν είχε ψηφιστεί με τέτοιο τρόπο στην Ολομέλεια έκθεση Γκρέκ δεν θα υπήρχε η νομοθεσία για την ενιαία αγορά. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ίσως να μπορέσουμε σήμερα να καταλήξουμε, αν και δεν πρόκειται για την τελική ψηφοφορία επί του θέματος. Θα ήθελα όμως και σήμερα η Επιτροπή μας να δείξει, να κάνει μια χειρονομία. Ξέρω λοιπόν Αντώνια, μας είπες ότι θα έχεις ορισμένες προφορικές τροπολογίες. Μην ξεχάσεις πότε ακριβώς πρέπει να ψηφιστούν. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε. Να συγκεντρωθείτε όλοι. οι εγκεκριθέντες, οι εμφαίνονται εδώ στον κατάλογο. Λοιπόν, θέλει και ο σκιώδης του ΕΛΚ, η σκιώδης του ΕΛΚ, με ένα σχόλιο, να μην αρχίσουμε γενική συζήτηση όμως. Όχι, δεν συνεχίζουμε τη συζήτηση, γιατί νομίζω όμως ότι είναι αργά τώρα για να ακουστούν το προφορικές τροπολογίες. Και των σοσιαλιστών είναι πάντοτε καθυστερημένες το θέμα είναι τόσο σημαντικό ώστε δεν αρκούν προφορικές τροπολογίες, χρειάζονται γραπτές. Αφού κάναμε τις συνεδριάσεις που είχαν προβλεφθεί. Πολλές φορές επιτεύχθηκαν όντως συμβιβασμοί και συμφωνήσαμε για πολύ σημαντικά σημεία. Όλο το θέμα είναι σημαντικό. Η κινητικότητα, ας πούμε, συμφωνήσαμε να είναι προτεραιότητα η αναγνώριση των επαγγελματικών της επαγγελματική κατάρτισης και προσόντων είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Η πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες, όλα αυτά, οι συντάξεις, Επιτέχθησαν, ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία, η επιτήρηση, η εποπτεία των αγορών, τα όργανα που ελέγχουν τις εισαγωγές και τώρα διαφωνούμε μόνο και μόνο για την κοινωνική πολιτική όπου προτείναμε κάτι που μπορεί τελικά να καταλήξει σε συμφωνία. Δείξτε κι εσείς λίγη καλή θέληση. Αφού πρόκειται για συμβιβασμό πρέπει και οι δύο πλευρές να υποχωρήσουν λίγο. Παρακαλώ να το αναγνωρίσετε αυτό και σήμερα καινούργιες τροπολογίες μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις νομίζω ότι είναι κάτι το τελείως ανάρμοστο. Καλά, ας μην ξαναρχίσουμε τη συζήτηση, αλλά πρέπει απλώς να ψηφίσουμε, αλλά ελπίζω και μετά την ψηφοφορία, αν παραμείνουν διαφωνίες, να λυθούν και αυτές μέχρι την Ολομέλεια. Λοιπόν, Υπότιτλος 1. Υπάρχουν εδώ αρκετές τροπολογίες. 33, 34, 35 και 36 όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Γι' αυτό περνάμε τώρα στην οίκον 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οίκον 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ή μάλλον όχι αποχές, αν κανείς ζητάει αποχές να το πει. Απασχόληση 1, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα για την ένα νέα με ολόκληρη σειρά τροπολογιών. Από ποια αρχίζουμε. 37 και 10 και 36 Άρχεται η ψηφοφορία επί των τριών αυτών τροπολογιών. Έληξε. Απορρίπτονται. Απασχόληση 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται καθώς και δύο άλλες. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτονται. Απασχόληση 9 δεν την ψηφίζουμε. Αναφορές 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 των αναφορών υπέρ. Κατά. Αποχές δεν το λέμε από Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Νομική 1. Άρχεται ηλεκτρονικά. Έληξε. Απορρίπτεται. Οι άλλες είναι δικαιοδοσίας άλλων επιτροπών. Συμβιβαστική 2 λοιπόν. Σε δύο τμήματα. όπως το ζήτησε το ΕΛΚ. Λοιπόν, το τμήμα 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Και τώρα ηλεκτρονικά για το τμήμα 2. Έληξε. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Τώρα 50 Α, όχι, όχι. Όχι 50. Συμβιβαστική 3 κατευθείαν. Συμβιβαστική 3. Άρχεται ηλεκτρονικά. Α, όχι, όχι, υπέρ, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Απασχόληση 2. Υπέρ κατά εγκρίνεται απασχόληση 3 υπέρ κατά εγκρίνεται λίμπε 13 υπέρ κατά εγκρίνεται 52 του Λουί Γκρέκ άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά έληξε εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Ναι, μας, το, μας είχαν προειδοποιήσει ότι θα υπάρχει μια τέτοια διαφορά, λοιπόν. Αναφορές 2, όχι. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 57. Άρχεται ηλεκτρονικά. Έληξε. Υπέρ. Ευχαριστώ. Η 58 καταπίπτει. 59 και νομική 16 μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οίκον 4 υπέρ κατά εγκρίνεται πώς επαλήθευση μάλιστα οίκον 4 ηλεκτρονικά έρχεται. έληξε α όχι απορρίπτεται Thank you, Mr. Kreutzmann. Uh... Ε, 18 19 λίμπε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα μια ολόκληρη σειρά καταπίπτει και πάμε στην στη νομική 13. Ναι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αναφορές 7 υπέρ. Αναφορές 7 ηλεκτρονικά. Έληξε. Εγκρίνεται. 19-17. Αναφορές 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αναφορές 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Αναφορές 10 νομίζω ηλεκτρονικά πρέπει ηλεκτρονικά. Ανάφ 10 άρχεται. Έλξε. Απορρίπτεται 17-20. Αναφορές 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Απασχόληση 2. Άρχεται ηλεκτρονικά. Έληξε. Απορρίπτεται. Απασχόληση 22. Δεν χρειάζεται εδώ να ψηφίσουμε. Είναι σχόλιο. Καθώς και της κυρίας Τούρουν είναι 72. 73 Μάντερς. Άρχεται ηλεκτρονικά. Έληξε. Εγκρίνεται. Περιφερειακή 15. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. ...76 και 75 μαζί υπέρ... ...κατά... ...εγκρίνεται... ...εγκρίνονται... ...η 74 κατά... 77 επίσης... ...78 επίσης... ...συμβιβαστική 6... Ο κύριος Γκρέκ θέλει να κάνει προφορική. Δέχεστε οι υπόλοιποι. Ναι. Ορίστε Λουί. Ναι, προφορική τροπολογία για να γεφυρώσουμε τις διαφορές μεταξύ των ομάδων. Να λέει, συμφωνεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 97 και το Χάρτων των θεμελιωδών δικαιωμάτων για να υπάρξει πιο ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία πρέπει η κοινωνική πολιτική να τεβεί στην καρδιά της πολιτικής μας και να συμβιβάσουμε την ανοιχτή οικονομία με βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση ενώ ταυτόχρονα θα εγγυάται τους κανόνες του ανταγωνισμού που δεν θα παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης και μεταξύ αυτών και τα εργασιακά, την κοινωνική νομοθεσία και ασφάλεια και τις συλλογικέ συμβάσεις όπως προβλέπει η χάρτα και οι συνθήκες. Καλεί την Κομισιόν να διασφαλίσει ότι με βάση τις προηγούμενες αξιολογήσεις μία ρήτρα κοινωνικής πολιτικής πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις πράξεις νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων και να είναι ορατότεροι αυτοί για να μπορούν οι πολίτες να έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στο σύστημα της εσωτερικής αγοράς. Τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ίση σημασία στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντολογική διάσταση των, της νομοθεσίας για κάθε νομοθέτημα της ενιαίας αγοράς έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σωστά η αξιολόγηση των τομέων και των διαστάσεων αυτών στη καθημερινή ζωή των πολιτών. Αυτή είναι πολύ ριζοσπαστική προφορική τροπολογία μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν την χώνεψαν όλοι καταλήλως. Νομίζω δεν πρόλαβε κανείς. θέλετε να ψηφίσουμε ως εναλλακτική στην 6 ή όχι, στη συμβιβαστική 6, γιατί εδώ είναι ολόκληρη νέα διατύπωση. Όχι, δεν. Σβάμπ. Κύριε Πρόεδρε, εμεί δεν είμαστε κατά των συμβιβασμών. Αλλά αυτό που μόλις προτάθηκε ήταν κάτι πολύ μακροσκελές και δεν το χωνέψαμε ακριβώς. Συμβιβασμός σημαίνει και κάποιες υποχωρήσεις ως προς την κοινωνική επίπτωση, όπως είπε επανειλημμένος το ΕΛΚ, αλλά για μας είναι δύσκολο να δεχτούμε αυτόν τον προφορικό συμβιβασμό σήμερα, σε αυτή τη φάση δηλαδή της διαδικασίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να εγκρίνουμε αυτή την προφορική τροπολογία σήμερα, διότι είναι πολύ αργά. Θέλετε να σας δοθεί κάποιος χρόνος να το σκεφτείτε, δηλαδή να διανεμηθεί γραπτός και να ψηφιστεί αργότερα ώστε να μπορείτε να έχετε το χρόνο να τη συζητήσετε λοιπά. Κρότσμαν. Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν παρόν όταν προσπαθήσαμε να πετύχουμε συμβιβασμό από αυτού. και είχαμε συμφωνήσει με το ΕΛΚ για διάφορα θέματα και τώρα τέτοιου είδους συμβιβαστική όπου να είναι προφορική και όχι γραπτή νομίζουμε ότι δεν είναι κάτι που μπορούμε να το, να το δεχτούμε. Έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια, κάναμε όλες τις προσπάθειες που ήταν δυνατές, έχουμε ξεπεράσει, έχουμε κάνει ήδη πολλές επαναχωρήσεις και δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Να ψηφίσουμε ό,τι είχε προταθεί. Δεν γίνεται αλλιώ. Καλά. Σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει πρώτα να γίνει αποδεκτός ένα συμβιβασμό πριν ψηφιστεί. Και φαίνεται ότι οι ομάδες δεν συμφωνούν γιατί δεν είχαν το χρόνο να το εξετάσουν. Μετά τη συνεδρίαση όμως πριν την Ολομέλεια μπορούμε να το ξαναδούμε. Κυρία Γκέμπχαρτ. Ευχαριστώ. Κάναμε όντως μεγάλες προσπάθειες και δεν καταλήξαμε στον συμβιβασμό αυτόν. Η ομάδα μας έκανε ό,τι μπορούσε για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό, δυστυχώς δεν επετέχθηκε. για λόγους που δεν καταλάβαμε πολύ καλά, δύο ομάδες ως προς την κοινωνική αξιολόγηση και την κοινωνική ρήτρα δεν συμφώνησαν. Θεωρούν ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και ότι η κοινωνική ρήτρα γίνεται δεκτή μεν, αλλά η αξιολόγηση για τις κοινωνικές επιπτώσεις είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Γι' αυτόν τον λόγο απορρίπτουμε την προφορική αυτή τροπολογία. Διότι οι φιλελεύθεροι και το ΕΛΚ δεν θέλουν ψηφοφορία. Ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα θα είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε καμία από τις τρεις εκθέσεις, γιατί χωρίς κοινωνική ρήτρα, που είναι τόσο σημαντική πτυχή, και το ανέφεραν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς την κοινωνική ρήτρα δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε καμία γνωμοδότηση. Στην Ολομέλεια λοιπόν μέχρι την Ολομέλεια πρέπει να το ξανασυζητήσουν οι ομάδες, αλλά όχι σήμερα να ακούγονται τέτοιοι προφορικοί συμβιβασμοί. Στο μέλλον θα συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες για να εγκριθεί αυτό που προβλέπεται για την κοινωνική ρήτρα και να υπάρξει συμβιβασμός. Μάλιστα, και εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή για να δούμε τι ακριβώς είναι η κοινωνική ρήτρα. Λοιπόν, περνάμε στον κατάλογο όσοι είχε. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 6. Έληξε. Απορρίπτηκε. 16-21. Τώρα πάμε στην τροπολογία 81 της κυρίας Ροζατούν και άλλων. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία είπα ηλεκτρονικά. Για την 81. Την 81. Αφού απορρίφθηκε ο συμβιβασμός. Έληξε. Αποδεκτή 81. Τώρα έχουμε πολλές που πίπτουν και πάμε στην παράγραφο 7.1 που είναι σειρά τροπολογιών διαγραφής που δεν καλυπτόταν από τη συμβιβαστική 6. Στη σελίδα 23 ε, έχω. 93, 94, 95, 96, 97. Άρχεται η ψηφοφορία για αυτές τις τροπολογίες. Άρχεται... για την διαγραφή του 7-1. Έληξε. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. 22 92 ηλεκτρονικά του Λουδοβίκου Γκρέκ. Έληξε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. και Εγκρίνεται και αυτή. Και τώρα η 93. για την 7, 7 η 93 PC1D για την εισαγωγικό τμήμα της παραγράφου 7. Έληξε Εγκρίνεται 27-10. 105 πέντε του Λουδοβίκου Γκρέκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται. Λίμπε 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Λίμπε 16 υπέρ κατά εγκρίνεται. Λίμπε 17 ηλεκτρονικά άρχεται. Έληξε. Απορρίπτεται. Βιομηχανία 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. 129 του Λουδοβίκου Γκρέκ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αναφορές 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Λίμπε και Νόμ 7. Στη σελίδα 32. Νόμ 7. Στην παράγραφο 9. Άι. Γιώτα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 139 της κυρίας Τούν και άλλων υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 142 Κρόιτσμαν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 199 καταπίπτει, απασχόληση 10 καταπίπτει. Τώρα στην παράγραφο 7.2 για τις βάρδιες. Πολλές τροπολογίες μαζί εδώ. Όλες μαζί λοιπόν για την παράγραφο 7.2 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός έληξε εγκρίνονται 21-15 ή 100 εκπίπτει απάσχ 14 Άρχεται η 100 απασχ 14 αρχεται η ψηφοφορια για την τροπολογία 14 πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται Έχουμε τώρα την τροπολογία 9 ε, της Τζούρι άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα έχουμε την τροπολογία 147. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Οίκον, 17 είναι προσθήκη, εγκρίνεται. 204 Αναμαρία, Μπάλα και άλλους, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Τώρα έχουμε την συμβιβαστική τροπολογία 12. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 158 που, που είναι στην σελίδα 40. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην συμβαστική τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβαστική τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα περνάω ε, στην τροπολογία 7 της ε, Επιτροπής Απασχόλησης. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ήμκο ε, 5. Με συγχωρείτε, διεθνούς εμπορίου, διεθνούς εμπορίου 5. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 14 ε, διεθνούς εμπορίου. 14 τε 14, πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 7 της Οικονομικής Επιτροπής, ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 18 της Οικονομικής Επιτροπής, άρχεται η ψηφοφορία για τη 18 της Οικονομικής Επιτροπής, πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 162. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, εγκρίνεται. 16 της οικονομικής ως προσθήκη, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην παράγραφο 11, 163 και 164 υπέρ, Άρχεται η ψηφοφορία 163-164 ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται με 22 υπέρ. 165-195 καταπίπτουν. 169 κατά. Εγκρίνεται. Οίκον 6 ως προσθήκη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Employment 23, απασχόληση 23, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 154, καλύπτεται από την οίκον 6. Περνάμε τώρα στην 170. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 170. Πέρα της ψηφοφορίας, εγκρίνεται, 25 προς 10. Τροπολογία 125, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 175. Άρχεται η ψηφοφορία για την 175. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 21-15 και 177-178 ε, εκπίπτουν. Περνάμε στο 182 του Λουί Γκρέκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 13 183 και 184 για διαγραφή. Άρχεται η ψηφοφορία για τις 183 και 184. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 21 προς 15. Αυτό σημαίνει ότι το 87, 186, 185 εκπίπτουν. Όχι, το 185 προτάθηκε. Και τώρα περνάμε ε, στην ε, συμβιβαστική τροπολογία 13. Ποιοι είναι υπέρ, Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε ε, στις άλλες τροπολογίες παρακολουθήστε με προσεκτικό. 13 απορρίφθηκε. Έχουμε τώρα ε, πρόταση jury 11. Τζούρι 11. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την Jury 11. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Οι άλλες τροπολογίες καταπίπτουν. Τώρα περνάμε ε, στην έξι της Επιτροπής Απασχόλησης. Χωρίς μικρόφωνο παρέμβαση. οι άλλες δεν έχουν γίνει, έχουν γίνει δεκτές. <clears throat> Έχετε δίκιο. We should now go through all of these votes. Έχετε δίκιο, ναι, ναι. Θα ψηφίσουμε για όλα αυτά. Με ονομαστική ψηφοφορία. ηλεκτρονική μάλλον. 15 της Επιτροπής Απασχόλησης, άρχεται η ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο γρήγορα παρακαλώ. συγχωρείτε. Πέρα της ψηφοφορίας, έχετε όλοι ψηφίσει τώρα. Απορρίπτεται. 188, άρχεται η ψηφοφορία. Α, 34. Μπορείτε να ψηφίζετε λίγο πιο γρήγορα, παρακαλώ. Απορρίπτεται. 10 της ΕΚΟΝ, Οικονομικής Επιτροπής, άρχεται η ψηφοφορία για την 10 της Οικονομικής Επιτροπής, πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται επίσης. Έχουμε την 6 της Επιτροπής Απασχόλησης για το τμήμα 1, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται επίσης. Έχουμε την 11 της ε, Επιτροπής Οικονομικής, πρέπει και για αυτήν να ψηφίσουμε, για την 11 της Οικονομικής Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται επίσης. Όλες αυτές οι τροπολογίες απορρίφθηκαν. Περνάμε λοιπόν τώρα στην τροπολογία 191 Άρχεται η ψηφοφορία για την 191. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με τον τρόπο αυτό, δεν ξέρω, αν θα ψηφίσουμε για την 119 ως προσθήκη όχι, την 192 ως προσθήκη. «192» για να είμαι σαφής. Ψηφίζουμε ως προσθήκη στην 191 που μόλις ε, υιοθετήσετε. Ψηφοφορία για την 192. Άρχεται η ψηφοφορία για την 192 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Έχουμε την 191 και συν την 192 ως προσθήκη. Αυτό σημαίνει ότι 194, 193 καταπίπτουν και περνάμε στο επόμενο φύλλο. Περνάμε τώρα στην 90. Την τροπολογία 90. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 90. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 207. Ναι, ναι. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 207. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται επίσης. Τώρα έχουμε χωριστή ψηφοφορία. Έχουμε δύο τροπολογίες, στην 200 και την 144, που είναι και οι δύο του κυρίου Κρότσμαν. Πώς ε, το κάνατε αυτό. Ζητήθηκε χωριστή ψηφοφορία, όπως αναφέρεται στον κατάλογο των ψηφοφοριών. Θα ψηφίσουμε λοιπόν Πρώτα απ' όλα για το πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται το πρώτο τμήμα και τώρα έχουμε μια άλλη τροπολογία για το τμήμα 2, άρχεται η ψηφοφορία για το τμήμα 2. 2. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται το τμήμα 2. Πρέπει να ψηφίσουμε επίσης για την Τζούρι 14. Ψηφίζουμε για την Τζούρι 14. Άρχεται η ψηφοφορία για την Τζούρι 14. πέρα στις ψηφοφορίες Απορρίπτεται επίσης. Τώρα λοιπόν περνάμε ε, στην ε, παράγραφο 7.3 και έχουμε ε, τις τροπολογίες 93, 94, 101. Άρχεται η ψηφοφορία για αυτές τις τροπολογίες. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνονται και συνεπώς η τροπολογία 102 και 103 καταπίπτουν. Τώρα περνάμε στην Ε, στην τροπολογία 198 De Jong, Evavits ε, για την ε, παράγραφο 17 για τις κοινωνικές κατοικίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 19 υπέρ κατά εγκρίνεται Συνεπώς έχουμε τώρα τις μεταφορές. Η 201 καταπίπτει. Περνάμε λοιπόν, σύμφωνα με τη γνώμη μου, στην τροπολογία 202. Συμφωνείτε όλοι, 202. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Χρειαζόμαστε Μπορούμε να αρχίσουμε την ψηφοφορία ηλεκτρονικά για τη 202. Πέρα στις ψηφοφορίας απορρίπτεται. Έχουμε λοιπόν τώρα ε, μια σειρά τροπολογιών της Επιτροπής Μεταφορών. Μπορούμε να ψηφίσουμε on block για όλες ε, τις ε, τροπολογίες. 4 έως 7 υπέρ κατά εγκρίνονται όλες. Ευχαριστώ τον συνάδελφο της Επιτροπής Μεταφορών. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 168. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 113 που είναι μια προσφύγη, ποιος ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Έχουμε τώρα την συμβιβαστική τροπολογία 14, ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 10 της Νομικής Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων στην σελίδα 58. Όχι, δεν ψηφίζουμε. Έχουμε 208 η επόμενη τροπολογία. Σωστά, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Έχουμε τη 12 της Επιτροπής Απασχόλησης, διότι έχουμε κάτι για το οποίο δεν ψηφίζουμε προηγουμένως. 12 της Επιτροπής Απασχόλησης, άρχεται η ψηφοφορία. 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 159. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 159. Για την ε, παράγραφο 16 γάμα απορρίπτεται 210. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 210. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τώρα έχουμε την τροπολογία 14 της ε, Περιφερειακής Επιτροπής. 14. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται ε, τροπολογία 8 της Επιτροπής Απασχόλησης, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας επίσης απορρίπτεται. Τώρα περνάμε ε, στην 5 της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 16 ε, θήτα, Α, υπάρχει καμιά αντίρρηση. Τη πέντε της ΛΥΜΠΕ. Περ, κατά, εγκρίνεται. Θα ε, βοηθούσα ο κύριο Σουάμπε. ε, μου έδειχνε πιο νωρί. Έχουμε την έξι της ΛΥΜΠΕ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Λίμπε 7. Όσοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται ε, πολιτικών ελευθεριών 8, 11, 12, 12 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα έχουμε ε, για υπότιτλο 4, 211, 212 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην συμβιβαστική ε, τροπολογία 15. Ποιοι είναι υπέρ. Χρειάζεται νομίζω ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμβιβαστική ε, τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά, εγκρίνεται. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 15. Περνάμε τώρα στο 247 ε, που είναι μετά από αρκετές σελίδες. Καλή δουλειά, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, ναι. Περνάμε τώρα στη 247. Κρέα κάμποσα που θεωρείται προσθήκη, προσθήκη στην συμβιβαστική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 247. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στη 227. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 243. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 247 που αντιστοιχεί στην ε, παράγραφο 17 σημείο θ, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται επίσης. Τώρα περνάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Συμβιβαστική τροπολογία 16, ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην ε, τροπολογία 9 της εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 17. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, τροπολογία 14 από την κυρία Τούρουναν και άλλος. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 14. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Έχουμε τώρα την ε, τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Enterprise 12, κυρία Πατρίτσια Τόια, Μαρκ Ταραμπέλα, πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται επίσης. Τώρα περνάμε ε, στην, στην συμβιβαστική τροπολογία 18, έτσι δεν είναι? Όσοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται Περνάμε στην συμβιβαστική τροπολογία 19 υπέρ κατά, επίσης εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, συμβιβαστική τροπολογία 20 όσοι είναι υπέρ κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην 29 ε, Σιμών Μπουζουτήλ υπέρ κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ χρειαζόμαστε ηλεκτρονική ψηφοφορία, νομίζω, για την τροπολογία 30. Πέρα τη ψηφοφορία Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 έχει καλυφθεί. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορία Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για την ε, τροπολογία 1. Πρώτη τροπολογία. Ψηφίζουμε για την πρώτη τροπολογία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται επίσης. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Νομίζω ότι Περατώθηκε αυτή η εργασία και αργότερα θα έχουμε την τελική ψηφοφορία. Θα έχουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών πριν από την ψηφοφορία για την έκθεση Μπουζόη. Μπορούμε να συνεχίσουμε τις ε, ψηφοφορίες μας. Η έκθεση Μπουζόη είναι η επόμενη έκθεσή μας. Είναι το κεφάλαιο για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Για να ξέρετε περί πρόκειται στην ε, πρόταση Αγαπητοί συνάδελφοι, επιχειρήν και μεγενθύνην. Δεν έχουμε εδώ πέρα κοινωνικές ρήτρες. Αυτά. Κύριε Μπουσόη, θέλετε να μας πείτε κάτι σε σχετικά. Πάρα πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Όλους τους σκιώδεις θέλω να ευχαριστήσω, το προσωπικό της Επιτροπής, τη Γραμματεία της ε, <clears throat> Επιτροπής, τους φιλελεύθερους. Θέλησαμε να έχουμε μια ευρεία υποστήριξη αυτής της έκθεσης και ήταν πολύ καλή συνεργασία και είμαι σίγουρος ότι η τελική απόλυξη θα είναι θετική. Ευχαριστώ πολύ τα μάλα. Καλά λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία λοιπόν για την έκθεση Μπουζόη. Τροπολογία 33. Μπουζόη. Ψήφι πέρα. Κατά. Δεκτή. Τζούρι 2. Ψήφι ηλεκτρονικά μάλλον για την Τζούρι 2. Πέρας. Απολύτως. 34 υπέρ, κατά, δεκτή. 35 σαν προστίκη. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. 37 δεν ψηφίζεται. 37. Και 12. Ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνει. 68 υπέρ κατά δεκτή. 39 Σφένσον υπέρ κατά απορρίπτεται. 41 υπέρ μάλλον ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 42 καλύπτεται. Ψήφι υπέρ 42 κατά δεκτή. Οίκον 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 45 υπέρ ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Είκον 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Είκον 3. Υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 17. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Απασχόληση 24. Υπέρ. Απασχόληση 24. Ναι, τα μπερδεύω και εγώ λιγάκι. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πέτη 4. Άρχεται η ψηφοφορία για την 4 ε, των αναφορών. Πέρας. Απορρίπτεται. Απασχόληση 4 ψήφι υπέρ. Μάλλον άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας είναι τα 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ζούρι 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. είναι τα 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Είναι τα 6. Διεθνές εμπόριο 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περιφερειακή 1. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περιφερειακή 5. Το αντίστοιχο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περιφερειακή 6. Ψήφι υπέρ. 6. Περιφερειακή είπα. Ηλεκτρονικά καλύτερα. Πέρας. απολύτερα 47 μπουζόι. Υπέρ. Κατά δεκτή. 48 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έχει απορριφθεί. 49 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτει. Ίντα 9. Ψήφι υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 1. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 58. Άρχεται η ψηφοφορία για την 58. Δεν έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία. Τώρα ξεκινάει. Πέρας. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Αν άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Συγγνώμη, εγκρίνεται. Πρέπει να συγκεντρωθώ λιγάκι. 61 εγκρίνεται, πάση περιπτώσει. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 18 τώρα. συγγνώμη, προηγουμένω. Η απασχόληση 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Σαν προσθήκη η απασχόληση 12. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστή 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 13 της βιομηχανίας. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αλλά ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. 13 βιομηχανίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Κύριε Σουάπ και κύριε Αγγέμπχαρτ, παρακαλώ κάντε το νεύμα σας προηγουμένως για να ξέρω. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 77. 74 τέσσερα μάλλον, συγγνώμη. Σαν προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Απασχόληση 13. Υπέρ. Κατά. <clears throat> Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με ισοψηφία. 78. Άρχεται η ψηφοφορία για την 78. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 και 79 δεν ψηφίσουμε. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περιφερειακή 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 89 Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 91. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 60. Ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 92 σαν προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Βιομηχανία 4. Το αντίστοιχο τμήμα είναι παράγραφος 9β. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περιφερειακή 13. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 107 και τζούρι 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 8 είπε. Άρχεται η ψηφοφορία στην ηλεκτρονικά για τη συμβαστική 8. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 87 Κρόιτσμαν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε εγκρίνεται με μία μονάχα διαφορά. Διεθνές εμπόριο 8. Άρχεται ψηφοφορία. Μάλλον υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. 1.33 Μπουζόι. υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οικονομική 7. Αρκετή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Οικονομική ενέα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Η, 10, η οικονομική δέκα. Τι ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ο κύριος Σφάμπ, χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο, κύριο Σφάμπ. Δεν ακούμε τον κύριο Σφάμπ. Νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε την ε, οικονομική 13, γιατί απερίφθη η οικονομική 10. Ψηφίσουμε την οικονομική 13. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 13. Καθυστερείται. Πέρας. Απορρίπτεται. Σαφώς. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 142. υπέρ κατά εγκρίνεται 86 <clears throat> Σούλη και άλλη, άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται συμβαστική 10 ψήφι υπέρ κατά εγκρίνεται Απασχόληση 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ω προσθήκη, περιφερειακή 2, το αντίστοιχο τμήμα. Ψήφι υπέρ, κατά, δεκτή. 144 <clears throat> υπέρ, κατά, Δεκτή. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 147. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 148. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 149 και 160. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 141-160. <clears throat> Πέρας εγκρίνεται. 151 ψήφι υπέρ κατά δεκτή. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 157 άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. 159. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Καλύπτουν οι υπόλοιπε. Συμβαστική 13. Υπέρ. Αυτή την ψηφοφορία για την συμβαστική 13. Πέρασε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Οικονομική 15. Έχει αλλάξει ο κατάλογος ψηφοφορίας, υπάρχει ένα πρόβλημα So, do you want me to read this out? This is a, an Econ 12. Αυτή είναι η οικονομική 12 που έχει συμφωνηθεί και νομίζω πρέπει να τη διαβάζω. Υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό της φορολογικής πολιτικής των κρατών μελών ώστε να μειωθούν τα φορολογικά εμπόδια στην ε, ενιαία αγορά και αντιμετώπιση της διπλής φορολογίας και του φορολογικού ανταγωνισμού. Αυτή είναι προστίκη για την οικονομική 12. Ψηφίζουμε λοιπόν αυτό το τμήμα με, ονομαστική, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κυρία Τούρουνεν, μπορείτε να το ξαναπείτε αυτό που είπατε. Πάρα πολύ γρήγορα τα είπατε νομίζω. Θέλετε να το ξαναδιαβάσω είναι ένα τμήμα της τροπολογίας οικονομικής 12, το οποίο πρέπει να προσταθεί στη συμβαστική τροπολογία. Τα ξαναλέω. Μπορείτε να κάνετε λίγη σιωπή να τα διαβάσω, παρακαλώ. Υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των εθνικών φορολογικών πολιτικών με τον στόχο να μειωθεί ακόμα περισσότερο το αριθμό των φορολογικών εμποδίων και προσκομμάτων στην εσωτερική αγορά και να αποφευθεί διπλή φορολογία και να αντιμετωπιστεί ο φορολογικός ανταγωνισμός. Κύριε Ζουβά, συγγνώμη πρόεδρε, δεν το καταλαβαίνω. Έχει εγκριθεί συμβαστική τροπολογία 13. Λέει ο κατάλληλος ψηφοφορίας ότι ακόμη και τροποποιημένη η 12 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Ο εισηγητής να μας εξηγήσει καλύτερα είχαμε καταρχήν αποφασίσει ότι καλύπτεται από την 13, αλλά ζητήθηκε το δεύτερο τμήμα, αυτό το οποίο διαβάσατε εσείς, να συμπεριληφθεί ως προστίκη, γιατί δεν καλύπτεται από τη συμβασική τροπολογία. Γι' αυτό δεν αναφέρεται στον κατάλογο ψηφοφορίας, γιατί αυτό αποφασίστηκε τελευταία τη στιγμή. Όποιος θέλει μπορεί να καταψηφίσει. Λοιπόν, λίγη σαφήνεια. Αυτό είναι κάτι που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. Και ζητείτε να το ψηφίσουμε και να το προσθέσουμε στη συμβαστική τροπολογία γιατί δεν καλύπτεται από την συμβαστική τροπολογία είναι στοιχείο ενός ψηφίσματος που έχει ήδη κατατεθεί. Και το ερώτημα είναι αν εγκρίνεται ή όχι για να ψηφιστεί και εγώ νομίζω ότι είναι παραδεκτό το ψηφισμό προς θήκη. Αυτό θέλει και ο εισηγητής εξάλλου. Δεν είναι ακριβώς το προφορική τροπολογία. Είναι κάτι που είχε υποβληθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία για την Οικονομική 12. Άρχεται η ψηφοφορία για αυτή την προσθήκη. Λίγο πιο γρήγορα παρακαλώ. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στην... Πού πάμε? Οικονομική 15. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 15. λέξεις. Απορρίπτεται. Ναι, λίγο πιο γρήγορα πρέπει να ψηφίσετε, λέει ο πρόεδρος. Δεν μπορώ να ξαναρχίσω την ψηφοφορία. Απορρίφθηκε, εν πάση περιπτώσει. Απασχόληση 16. Υπέρ. Κατά. Λοιπόν, πάλι, απασχόληση 16. Άρχεται. Λήξεις. Απορρίπτεται. Απασχόληση 18. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 169, <clears throat> άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Διεθνές εμπόριο 10, το αντίστοιχο τμήμα, για την παράγραφο 16β. Άρχεται ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Με ισοψηφία. Καταλογνων8 Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Είναι τα 11 διεθνές εμπορίο 11, αρχιέται ψηφοφορία. Λήξεις. Απορρίπτεται. Διεθνές εμπόριο 12. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Διεθνές εμπόριο 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 180 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 181 άρχεται την ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 187 άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Νομική 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Απασχόληση 9 ως προσθήκη για την ε, προηγούμενη άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. <clears throat> Απορρίπτεται. 189 του εισηγητή υπέρ κατά δεκτή 91 άρχεται η ψηφοφορία 191 αν πέρας απορρίπτεται 192 άρχεται όχι συγγνώμη 192 ψήφι υπέρ κατά δεκτή 193 είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές δεν κρίνεται. 194 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 195 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15. Κύριε Σουάμπ, βλέπετε αρνητικά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Πάμε στην τροπολογία 200. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 201 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 202 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 214 που είναι διαγραφή, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Εκπίπτουν οι υπόλοιπε τροπολογίε. Πάμε στην 220, πάλι για διαγραφή. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 221 κροτσμαν υπέρ, δεκτή. Ήτρε ένα σαν προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περιφερειακή 7, 8 και 9 μπορούμε να τις ψηφίσουμε. Όχι, δε. Περιφερειακή 7. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Περιφερειακή 8, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περιφερειακή 9, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Πάμε στην παράγραφο 22. Η τροπολογία ζουβά σε δύο τμήματα. Για να ελέγξουμε τώρα τι έχει γίνει. Το πρώτο τμήμα, μόνο πρέπει να ψηφίσουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δύο 23. Ψήφι. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δύο Δεν μετακινήθηκε. Την ψηφίσουμε, εν πάση περιπτώσει. Έρχεται η ψηφοφορία για τη 225. απορρίπτεται. 226 όχι δεν την ψηφίζουμε. 27 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 190 εκπίπτει. Συμβαστική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Ε, ηλεκτρονικά. Άρχεται την ψηφοφορία για την 17. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 230 του εισηγητή. Ψήφι υπέρ. πέρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 2.31. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίφθηκε. Απασχόληση 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Νομική 5. Ε, ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις πια. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Δεν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. <clears throat> Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Εντρίνεται. Δεν ψηφίζουμε τα επόμενα. Έχουν μεταφερθεί. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία στις 13. Πέρασε. Απορρίπτεται. 14 ψηφίζουμε Άσχετη ψηφοφορία. Πέρας. Ε, απορρίπτεται. Η Οικονομική Επιτροπή D ψήφι υπέρ κατά δεκτή τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 18 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 ψήφι υπέρ κατά εγκρίνεται. 21 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται 22 άρχεται η ψηφοφορία για την 22 πέρας απορρίπτεται 23 άρχεται η ψηφοφορία ναι πέρας εγκρίνεται 24 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 27. 26 δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. 27 ψήφι πέρα Κατά. Εγκρίνεται. 28. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 29. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 30. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξεις. Απορρίπτεται 31. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εντάξει, απολύτω. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε τις τελικές ψηφοφορίες ε, των τριών εκθέσεων ηλεκτρονικά. Θέλετε να πείτε κάτι πρώτη, πρώτου κάνουμε την τελική ψηφοφορία, κύριε Γκέμπχαρτ. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους ε, τρεις συζητητές για το έργο τους. Έχουν γίνει πάρα πολλά και πάρα πολύ θετικά πράγματα τα οποία τα έχουμε ψηφίσει. Αλλά πρέπει κατά τα άλλα να σας υπενθυμίσω ότι είναι ορισμένα σημεία που έχουν να κάνουν με την κοινωνική διάσταση της ε, εσωτερικής αγοράς έχουν καταψηφιστεί με την συμμετοχή των φιλελευθέρων. Αυτό σημαίνει σε τελική ανάλυση ότι η ενία αγορά έχει πια μονάχα ένα οικονομικό και χρηματοοικονομικό στοιχείο, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να είναι στο κέντρο της νομοθεσίας δεν μπορούν να καλυφθούν. <clears throat> Αυτό κάνει για μας αδύνατο να ψηφίσουμε ως πολιτική ομάδα θετικά υπέρ των τριών αυτών εκθέσεων. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Γιατί υπολείπεται πάρα πολύ αυτό το περιεχόμενο σήμερα από αυτό που είχαμε αποφασίσει στην έκθεση Louis Grech. Και υπολείπεται επίσης πάρα πολύ σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε ψηφίσει στην έκθεση Μπερές της Επιτροπής Κρίσης. Μας κάνει λοιπόν αδύνατο να υπερψηφίσουμε, γιατί υπολείπεται ακόμα και σε ορισμένα σημεία από αυτό το οποίο είχε προτείνει η ίδια η Εκτελεστική Επιτροπή. Λοιπόν, για μας είναι <clears throat> απόλυτα ανεύθυνο να πούμε εμεί ω βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι υποστηρίζουμε και εξυπηρετούμε του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο η πολιτική μου ομάδα θα αναγκαστεί να καταψηφίσει και τι τρει, μάλλον να κρατήσει στάση αποχής για τι τρει αυτέ εκθέσει, γιατί δεν μπορεί να τι υπερψηφίσει. Η αποχή μα δείχνει ότι εμεί έχουμε τη θέληση μαζί με όλες τις άλλε πολιτικές ομάδες να συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει και τι επαφέ, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να ενσωματώσουμε όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ρήτρα, όπως είναι τα θέματα της ε, απόσπασης χάρη εργαζομένων, όπως είναι τα θέματα τα οποία άπτονται των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, σε ό,τι αφορά επίσης τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρία Κανιέτε, έχουμε ακόμα να κάνουμε πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Για όλους αυτούς τους τομείς Πιστεύω ότι χρειάζεται μια περαιτέρω διαβούλευση μεταξύ των ομάδων, ώστε να μπορέσουμε στην Ολομέλεια να καταλήξουμε σε μια ψηφοφορία και σε μια κοινή θέση, η οποία θα έχει θετικό αποτέλεσμα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς δεν θα έχει θετικό περιεχόμενο και εγώ επομένως ζητώ από την πολιτική μου ομάδα να κρατήσει στάση αποχής και για τις τρεις αυτές εκθέσεις, ώστε να κρατήσουμε ανοιχτή την πόρτα για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και να μπορέσουμε ενδεχομένως να καταλήξουμε σε λογικές συμβαστικές λύσεις ενώ ολομέλης. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Ίσως οι άλλες πολιτικές ομάδες αν θέλουν να κάνουν κάποιο σύντομο σχόλιο για τα θέματα αυτά γιατί είναι 12 και 4 και πρέπει να κάνουμε την τελική ψηφοφορία. Κύριε Σφάπ και κύριε Κρότσμαν, κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν ξέρω αν κυρία Ρούλα θέλει να λάβει το λόγο. Κύριε Σφάπ, <clears throat> σας ευχαριστώ πρόεδρε. εγώ νομίζω ότι είναι για μας απόλυτα ανεύθυνο η σοσιαλιστική ομάδα να θέλει να θέσει πίεση τώρα στα άλλα πολιτικά κόμματα γιατί δεν ακολούθησαν κατά 100% αυτά τα οποία θέλαν οι σοσιαλδημοκρατές. Εμείς ακολουθήσαμε την έκθεση Λουί Γκρέχ ε, η οποία υποστηρίχθηκε από όλους γιατί τώρα δεν το δέχονται αυτό οι σοσιαλιστές, δεν ξέρω. Επίσης η κοινωνική λύτρα υπάρχει εδώ, ε. εγώ δεν νομίζω ότι δεν είναι ισορροπημένη από κοινωνική άποψη έκθεση. Αυτό το απορρίπτω με τρίτον σαν ΕΛΚ. Εμεί θελήσαμε να έχουμε μία έκθεση. Οι σοσιαλιστέ είπαν όχι, θα κάνουμε τρει εκθέσει. Τώρα δεν είναι λογικό να κρατήσουν μια θέση χωριστά ε, από κοινού κατά των τριών εκθέσεων. Γιατί αυτοί είπαν ότι είχαν προβλήματα σε μία έκθεση μονάχα και όχι στι άλλε. Εμεί θέλουμε να προχωρήσει η πράξη αυτή για του πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κοινωνικά δικαιώματά του σε επίπεδο εσωτερική αγορά λένε ότι η αποχή τους ανοίγει τη δυνατότητα για μια συμβαστική θέση, αλλά εγώ νομίζω ότι αντίθετα έχουμε καταφέρει σήμερα να εγκρίνουμε πολύ καλές εκθέσεις και δεν νομίζω ότι χρειάζεται μια περαιτέρω τέτοια διαπραγμάτευση. Κρότσμαν. Κρότσμαν. Εγώ εκφράζω και εγώ τη λύπη μου για αυτά τα οποία είπε η κυρία Γκέπχαρτ. Εμεί έχουμε προσπαθήσει σε πάρα πολλέ συζητήσει η έκθεση Korea the Campus να μπορέσει να αντιμετωπίσει πλήρω και συγκεκριμένα όλα τα κοινωνικά αυτά θέματα για του πολιτέ της Ευρώπης. Εμείς προχωρήσαμε, αλλά εσεί κυρία Γκέπχαρτ έχετε επιμείνει πάντα σε αυτή την εφελώδη κοινωνική ρήτρα. εμεί είπαμε να έχουμε συγκεκριμένε αντιμετωπίσει προβλημάτων και αναγκών όταν υπάρχουν. Ήμασταν έτοιμοι να το πράξουμε αυτό και <clears throat> ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε εσείς να το αντιμετωπίσετε με ένα ναι ή με ένα όχι. Εμείς κάναμε προσπάθειες να καλύψουμε τις ανησυχίες σας, γιατί και εμείς θέλουμε μια κοινωνική Ευρώπη. Έχουμε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς και αυτή είναι η έννοια η οποία καλύπτει την ευρωπαϊκή αγορά και έχουμε προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή, κυρία Γκέπχαρτ. αν υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη τα οποία δέχονται τη συναπόφαση εργαζομένων και εργοδοτών όπω γίνεται στη Γερμανία, πολλά από τα προβλήματα τη εσωτερική αγορά θα, θα είχαν λυθεί. Δεν μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την κοινωνική αυτή ρήτρα σαν μια γενική ε, αιτία απόρριψη ή αποχή. Κυρία Γκέπχα, θα, θα σα παρακαλούσα να είστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτά τα οποία ζητάτε. Καταλαβαίνω τα σχόλια των μέλων της ομάδας σας. Ε, κυρία Ρούλα. Ούτε και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας για την έκθεση Κάμπους. Θα καταψηφίσουμε την έκθεση Κορέαντα Κάμπους για ένα απλό λόγο. Με την απόφαση αυτή θα, πρέπει, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο βλέπουν οι πολίτες μας σαν έλλειμμα στον ε, κοινωνικό τομέα, συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και ενδιαφέροντος. Περιμένουμε εδώ, εδώ οι πολίτε να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία από την κοινωνική αγορά. Φοβούνται ότι οι υπηρεσίε αυτέ γενικού ενδιαφέροντο θα βρεθούν κάτω από μεγάλη πίεση λόγω τη ρύθμιση τη εσωτερική αγορά. Η απόφασή μα κατά τη έκθεση κάμπου δεν προσδιορίζει τη θέση μα για τι άλλε δύο εκθέσει και δεν ακολουθούμε την κυρία Γκέπχαρτ. Εμεί υποστηρίζουμε την έκθεση Καλνιέτη και την έκθεση Μπουζόη, γιατί έχουν επιτευχθεί πολύ καλέ συμβιβαστικέ λύσει και εμεί θεωρούμε ότι μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με την έκθεση Μπουζόη και επομένως μπορούμε να την υποστηρίξουμε και να την προχωρήσουμε. Κατά τα άλλα, κάνουμε μια έκκληση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάνουμε μια έκκληση για τις άλλες πολιτικές ομάδες να υπάρξει και πάλι μια διαβούλευση πριν από, τις, ε, πριν από την Ολομέλεια, γιατί για τα θέματα της Ευρώπης των ε, ε, την κοινωνική Ευρώπη, την Ευρώπη των πολιτών στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει να βρούμε μια λύση στην έκθεση Κορέα Campus που να αντιμετωπίζει την προστασία των πολιτών και την προστασία των υπηρεσιών γενικού συμφέροντο και ενδιαφέροντο. Αυτό θα ήταν και η ευχή μα να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση για όλα αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι ο κύριος Φόξ είναι ο επόμενος. Έναν από κάθε ομάδα και μετά θα κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για τρεις καλές εκθέσεις και θέλουμε να ευχαριστήσουμε από την ομάδα μας την, ε, τις, ε, τους ε, εισηγητές αυτά που είπε. Είναι σημαντικό σημαντική εργασία η οποία συμπληρώνει την ενιαία αγορά και θα ε, φέρει ευημερία στους πολίτες, ε, την καλύτερη προστασία που μπορούμε να προσφέρουμε στα άτομα ή να τους προσφέρουμε απασχόληση και υπάρχει ε, κίνδυνος αν αυξηθεί το κόστος ή οι δαπάνες πάρα πολύ, που ορισμένοι δεν θα έχουν δουλειά, πάρα πολλά άτομα θα είναι άνεργοι, γι' αυτό θα ήθελα να κάνω έκκληση να ψηφίσετε υπέρ των εκθέσεων αυτών. Τους ε, τρεις ε, ραπορτές, Ωστόσο, θεωρούμε ότι όπως έχουν διαμορφωθεί οι εκθέσεις σήμερα, δεν περιλαμβάνεται πλέον η ισοζυγισμένη προσέγγιση για τις δράσεις που θα θέλαμε να καλέσουμε την Κομισιόν να αναλάβει. Μας φαίνεται ότι αρκούμαστε μόνο στο να επικροτούμε τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την Κομισιόν. Γι' αυτό εμείς θα απόσχουμε. Ευχαριστώ. Okay. Πολύ καλά. Δεν θα, θα πόσχεται και για τις τρεις εκθέσεις και στις τρεις εκθέσεις. Πολύ καλά. Νομίζω ότι είχαμε μια συζήτηση και έλαβαν το λόγο όσοι ήθελαν, όσα μέλη ήθελαν. Δεν θα ήθελα να προχωρήσουμε περαιτέρω στη συζήτηση. Κύριε Σβάμπ, πρόκειται για ένα διαδικαστικό ή θέλετε να ξανανοίξετε τη συζήτηση. Α, είναι για... Θέλετε να μιλήσετε ή ψηφίζετε θα πάρουμε λοιπόν ε, χωριστά, θα ήθελα, πρωτού περάσουμε στην ε, ψηφοφορία, εγώ ως πρόεδρος, θα ήθελα πρώτα απ' όλο να ευχαριστήσω όσους ε, συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Είδατε τον αριθμό των μελών και είδατε πόσο σε βραχή χρονικό διάστημα έγιναν όλα αυτά. Και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και άλλες επιτροπές οι οποίες συνέβαλαν σε αυτή την εργασία και χαίρομαι που πήγε τόσο καλά αυτή η εργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ηγητές για αυτή τη δέσμευση ε, και την συνεργασία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, μπορούν να συνεργαστούν εύκολα και απλά οι επιτροπές χωρίς να έχουμε ε, τον κανόνα 50 κλπ. Νομίζω ότι η καλή σύμπραξη, η καλή ε, συνεργασία, η αγαστή συνεργασία είναι κάτι που μας δείχνει πώς μπορούν να συνεργαστούν μέλη, αναπληρωτικά μέλη των επιτροπών μεταξύ τους. Όπως είπα στην αρχή, λυπούμε που δεν μπορούμε Ε, σήμερα ε, να υιοθετήσουμε ε, χωρίς κανένα χαρακτηρισμό αυτές τις τρεις εισηγήσεις όπως είπε η κυρία Γκέμπαρτ και ο κύριος Σβάμπ έχουμε άλλη έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε πριν από την τελική ψηφοφορία και δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε για την πράξη για την ενιαία αγορά εκτός αν έχουμε υιοθετήσει τη εισήγηση και νομίζω ότι αυτή η εισήγηση έδωσε ένα σαφές μήνυμα ε, διότι ήταν η ενιαία αγορά για τους καταναλωτές και τους πολίτες και όλες οι πολιτικές ομάδες ε, την υποστήριξαν. Αν λοιπόν βασιστούμε σε αυτό σημείο κίνησης, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία αρκετά γρήγορα, διότι δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Πρέπει λοιπόν να συμπληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε την ενιαία αγορά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και οικονομική μεγέθυνση. Νομίζω ότι το ΕΛΚΑ, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες και όλες οι ομάδες θα πρέπει να δουν αν μπορούμε να κάνουμε πρόοδο όπως είχαμε κάνει με την αρχική εισήγηση Λεγκρέκα. Και τέλος ξέρω ότι υπήρξαν συζητήσεις για τη δομή, τη διάρθρωση των όσων κάναμε. Θα ήθελα να σας πω ότι η όγκος ε, της εργασίας ε, των εισηγητών δικαιολογεί την απόφασή σας να έχουμε τρεις χωριστές εισηγήσεις, διότι σε αυτές τις προτάσεις είχαμε τόσα πολλά θέματα, θα μπορούσαμε λεπτομερώς να καλύψουμε όλα αυτά τα θέματα. Γι' αυτό ήταν καλό που είχαμε τρεις εισηγήσεις. Αυτό ε, το συμβουλεύω και σε άλλες επιτροπές όταν έχουν να κάνουν με λεπτομερείς και ενδελεχείς προτάσεις. Δεν μπορεί μία εισήγηση να καλύψει ένα τόσο ευρύ θέμα. Αυτό είναι κάτι που θα το λάβω υπόψη και για τους Πρόεδρους των Επιτροπών, διότι ε, θα έχουμε πολλές από αυτές τις μεγάλες ε, πρωτοβουλίες ε, στις οποίες θα περιλαμβάνεται η εργασία πολλών επιτροπών. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά για κάθε εισήγηση. Πρώτα απ' όλα έχουμε την εισήγηση Καρνιέτη για την διακυβέρνηση ε, πρόκειται ε, για την τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την εισήγηση Καρνιέτη. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 37 υπέρ, ε, μία ψήφο κατά και 12 αποχές. Τώρα τελική ψηφοφορία για την εισήγηση ε, του καθηγητή Αντώνιο Φερνάντο Κορέια Ντεκάμπος ε, για την ενία αγορά για τους Ευρωπαίους. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 21 υπέρ, 3 κατά και 13 αποχές. Και τέλος ε, η εισήγηση Κριστιαν Μπουζόη για την ενή αγορά για επιχειρήσεις και ανάπτυξη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Επίσης εγκρίνεται με 24 υπέρ, καμία ψήφο και 13 αποχές. Σας ευχαριστώ όλους, σας υπενθυμίζω ότι σήμερα ε, το απόγευμα η συνεδρίαση είναι σε άλλη αίθουσα, στην αιθουσα 66 6Q2. Έχουμε ένα, μια, επίσης μια συνεδρίαση για εναλλακτική